Liebe Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν, θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα. Βλέπω ότι έχουμε αποδεκατιστεί άλλωστε. Πραγματικά οι τελευταίες δυόμιση ώρες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, έγινε μια πολύ καλή συζήτηση με εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες που με πολύ μεγάλη σαφήνεια μας είπαν τις δικές τους απόψεις. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε και να συζητήσουμε επί όλα αυτά τα θέματα, αλλά τυπικά πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν την ε, έκθεση αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω σύντομα το λόγο στην ε, Χέλγα Τρούπελ. Δεν ξέρω αν έχει και να προσθέσει κάτι σε σχέση με τα όσα είπε ε, πριν από λίγο, αλλά παρόλα αυτά έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πράγματι η εκρόση αυτή ήταν ε, πάρα πολύ καλή, ε, με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές εχμές από τη δική μας πλευρά. Ιδίω αυτά που είπες εσύ, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων, αλλά δεν θέλουμε να μπλέξουμε τα διάφορα προγράμματα. Να δοθούν περισσότερα χρήματα για την εγγύηση για την νεολαία, και ταυτόχρονα να υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός όσον αφορά την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό και ξεχωριστά χρήματα, ξεχωριστή χρηματοδότηση βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στόχο που δεν έρχεται σε αντίθεση και με του στόχου τη Κομισιόν. Θέλουν και εκείνοι να ενισχυθεί ο εθελοντισμό και η αλληλεγγύη και ταυτόχρονα θέλουν και εκείνοι να ε, αντιμετωπιστεί η νεανική ανεργία. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε όλα στην ακρόαση. Αυτό που με ενδιαφέρει ε, θα ήταν να ακούσω ε, απόψεις ε, συναδέλφων ε, που ίσως δεν έχουν ακούσει. Νομίζω ότι με εξαίρεση τον Έλληνα κομμουνιστή και τους ακροδεξιούς όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να συμφωνήσουμε, να βρούμε συνένεση Νομίζω ότι αυτό που θα μας απασχολήσει ιδίω είναι το περιεχόμενο του Erasmus ε, Plus, αν θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό προγράμματα που θα σχετίζονται περισσότερο με την απασχόληση. Θα με ενδιέφερε να ακούσω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων. Έχουμε υπόψη μας βεβαίως τι ε, συζητήσεις ε, βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το θέμα αυτό και στο Συμβούλιο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω απλώς ότι η προθεσμία για την καταβολή τροπολογιών είναι η 20 Οκτωβρίου και ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου. Δυστυχώς αναβλήθηκε η ψηφοφορία μας διότι ε, αν είχαμε ακολουθήσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αποσχόλησης θα ε, ήταν, θα γινόταν πολύ άμεσα πριν από τη δική μας ψηφοφορία και λόγω του ειδικού βάρους που έχει η Επιτροπή Απασχόλησης σε αυτό το θέμα θελήσαμε να ε, ε, αφήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Βάσει του άρθρου 54 η Επιτροπή Απασχόλησης είναι συνδεδεμένη επιτροπή. Ταυτόχρονα έχουμε και επιτροπές Ρέτζι, ε, Άγκρι ε, που θα γνωμοδοτήσουν ε, για αυτήν την έκθεση. Είναι η Επιτροπή Απασχόλησης σίγουρα παίρνει στα σοβαρά αυτήν την έκθεσή μας. Γι' αυτό και είπαμε να γίνει η ψηφοφορία στις 20 Ιανουαρίου. Τρεις ανθρώπους έχω στο κατάλογο μιλητών αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μετά από αυτό ε, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και την σημερινή συζήτηση. κυρία Σόντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την ακρόαση, διότι οι φορές ήταν έξοχες. Όλα όσα ακούσαμε επί του θέματος ήταν χρησιμότατα για μας και για τις μεταγενέστερες εργασίες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξίσου την Χέλγα Τρίπελ για το σχέδιο εκθέσεώς της, που καταδεικνύει σαφώς κατά την άποψή μου με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Υποστηρίζω πλήρως το σχέδιο αυτό της αλλαγής του τίτλου, την πρώτη αλλαγή του τίτλου. Και θα ήθελα να πω ότι το αρχικό σχέδιο κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ένα σημαντικό, μια σημαντική έλλειψη. Αν δείτε τους στόχους του κανονισμού που προτείνει όσον αφορά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στους συγκεκριμένους στόχους και στους γενικούς στόχους δεν βλέπετε τη λέξη εθελοντισμός. Η λέξη εθελοντισμός δεν ανήκει στους στόχους ε, του σώματος αλληλεγγύης. Εδώ δεν πρόκειται για μια επίσημη ε, φιλοδοξία, ίσως να δείχνει κάτι. Η κατεύθυνση της εκθέσεως της Helga Triple θα απαιτήσει να εστιαστούμε και από αυτού του τμήματος. Συμφωνώ απόλυτα με διάφορες προτάσεις που μας παρουσιάζει και αν μειώναμε την πτυχή της απασχολησιμότητας, αν αυτό το τμήμα διαγραφόταν, εν τη αυτή περιπτώσει αυτό θα μπορούσε να παραμείνει στα πλαίσια του Erasmus Plus. Και θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο την αλληλεγγύη, τον οθελοντισμό και θα ήταν πράγματι αυτή μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα στον τομέα. Απ' την άλλη θα πρέπει να απαιτήσουμε ότι στο θέμα της απασχολησιμότητας να τονίσουμε και να ισχύσουμε την αλληλεγγύη. Αυτό ανήκει σε άλλα προγράμματα διαφορετικά. Θεωρητικά ότι αυτό το σχέδιο είναι πάρα πολύ λογικό, θα πρέπει να τύχει υποστηρίξεως. Αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Σας και όδηση συγγήτρια. Περιμένω με ανυπομονησία τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα. Λοιπόν, πράγματα που δεν είπαμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όσον αφορά το τίτλο, το όνομα, εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Από την αρχή είπα ότι δεν είναι πραγματικό σώμα. Δεν υπάρχει ε, νομικό πρόσωπο που να αποκαλείται σώμα. Η μόνιμη ανησυχία είναι χρησιμοποιείται η λέξη σώμα ήδη. Ε, το έχουν ζήσει όμως κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχει αυτό και κυκλοφορεί σαν ονομασία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι ε, υπάρχει αυτή η προπτική με αυτόν τον τίτλο. Να πούμε απλώς πρωτοβουλία. Μίσος είναι κάπως περιορισμένο, μειώνει την εμβέλεια. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Θέτω το πρόβλημα. Δεύτερον, ο δρόμος που σκεγγραφήθηκε και από την υποφαινόμενη όταν προσπαθούσα να εξηγήσω και στην Επιτροπή Απασχόληση το θέμα της απασχόλησης είναι απασχολησιμότητα, κατάρτιση, όχι απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Και μπορούμε να βάλουμε και την εγγύηση για του νέου εκεί αυτή η σαφήνεια ότι στόχος, όπως έλεγε και η κυρία Σοϊντράβα, είναι εθελοντισμός για λόγους αλληλεγγύης και για σκοπούς αλληλεγγύης, πρέπει να παραμείνει αυτό βασικός προσανατολισμός. Αυτό που απορρέει και από την άριστη έκθεση και συγχαρητήρια για την έκθεση, για τη μελέτη μάλλον, είναι άλλο θέμα της διαμεσολάβησης που αφήνεται εκτός, διότι είναι άμεση η σχέση μεταξύ του νέου και της ένωσης του φορέα αυτό που υπήρχε πριν λείπει. Φορείς διαβούλευσης λείπουν και ο ρόλος των δικτύων. Ρωτώ κάτι από την Έλγα. Στο κείμενό σου που αφορά την ενδιάμεση οργάνωση, οργανώσεις ενδιάμεσης, εκεί αναφέρεσαι σε αυτό, δηλαδή οργανώσεις, youth forum κλπ. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεσαι στα δίκτυα που υπάρχουν και βοηθούν. Εντάξει, ωραία, Ωραία, λοιπόν. Συμφωνώ. Όμως ίσω θα ήταν χρήσιμο αυτά να αποκληθούν σαν οργανισμοί διαβούλευση σε συγκεκριμένες περιόδους και τόπους που κάνουν επαλήθευση τη ποιότητα. Δεν μπορούμε να δώσουμε το ίδιο σήμα. Εγώ δεν θέλω να μπει ιδιωτικό στο μέσο εδώ. Πιστεύω ότι θα προκαλέσει σύγχυση. Ίσως μπορούμε να πούμε επιχειρήσεις που είναι φιλικές, ε, συνεργάζονται με το σώμα αλληλεγγύης θα, θα το ψάξουμε. Να εξετάσουμε τους πόρους και λοιπά ποιοι συμμετάχουν. Δεν είναι εκείνοι που απασχολούν και προσλαμβάνουν τους εθελοντές. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια. Αυτό είναι το σημαντικό, δεν προσθέτω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντάχει και εγώ θεωρώ ότι με σαφήνεια διαφάνει η απέτηση και ανάγκη να αποφύγουμε λήψεις μεταξύ των διαφόρων ζητημάτων και αν υπάρχουν επικαλύψεις δεν υπάρχει σαφήνεια. Άρα θα έχουμε έναν κανονισμό που τίθεται μέσα σε ισχύ που θα είναι Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτή την πλευρά λοιπόν. Λοιπόν, τα διάφορα ε, προβλήματα που πιστώθηκαν μας οδηγούν να αποφύγουμε κάτω από το ίδιο πλαίσιο να υπάρχει κάτι που σχετίζεται με την εργασία, εργασία απασχόληση ακόμα και αν είναι κακοπληρωμένη και από την άλλη πλευρά μια προσέγγιση αφορά τον εθελοντισμό που δεν αποσαφηνίζει κάτι σημαντικό ότι υπάρχει ο δωρεάν χαρακτήρας της υπηρεσίας αν αυτό δεν τονιθεί κάτω από την αιγίδα τη γενική μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Τα υπόλοιπα σαφώς τονιστήκαν. Ε, όσον αφορά αυτή την πτυχή, όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, για να φτάσουμε στον εθελοντισμό, όπως αναφέρθηκε, αναφέροντα το άθρο 2 τη συνθήκη τη Ένωση, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει μια διευκρίνηση, μια παραπομπή και στο προήμιο. Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει μια παραπομπή, μια αναφορά. Το λέω με αναφορά στο εξή ότι αυτή η πτυχή της αλληλεγγύης, αλληλεγγύης, αλληλεγγύης είναι μία από τις έννοιες, από τις κοινέ αξίες που όχι τυχαία συνεχώς επικαλούμεθα, που διαχωρίζεται από όλα τα άλλα. Πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αναφέρεται. Ίσως μπορούμε περαιτέρω να το τονίσουμε αυτό και να το αξιοποιήσουμε στα πλαίσια της σαφήνειας. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα μπορούσα να τα προτείνω στον αφορά τον καθορισμό του όλου ο κανονισμό, θέλω να καταλάβω. Ποιο είναι οι οργανισμοί αποστολή και υποδοχή, αν θέλετε. Ακολουθείτε Μία πτυχή μεταξύ άλλων που πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθεί. Επειδή είναι ο κανονισμο θέλω να καταλάβω ποιοι είναι οι, οι οργανισμοί ε, αποστολής και υποδοχής αν θέλετε. Απο, ε, ακολουθείτε μια διαδρομή, δύο εβδομάδες, δύο μήνες κλπ. Δεν θα πρέπει να παραμείνει αόριστο αυτό. Αλλιώς φοβάμαι ότι αυτό το σχέδιο κειμένου, αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το πρόγραμμα που θα μπορούσε να είναι κάτι που έχει σωστό μέλλον, να χρηματοδοτηθεί σωστά, μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα φάρος πραγματικά πρότυπο. Αλλά αν τελικά ε, εάν τελικά δεν τονιστούν και ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε μια εσόριξη, μια κατάρρευση του όλου προγράμματος. Λοιπόν, θα πρέπει αφού βρούμε τα προβλήματα να βρούμε και τις απαντήσεις. Και νομίζω ότι το βασικό μήνυμα που απέρευσε και διαφάνει είναι η σαφήνεια και αυτό πρέπει να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει το λόγο. Μόνο αν θέλετε, μόνο αν θέλετε. Δεν πιέζουμε κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ε, το ότι ήταν πολύ χρήσιμο που καθίσαμε και ακούσαμε τους εμπειρογνώμονες. Ε, έχουμε κάνει ένα σωρό σημειώσεις ε, με τα όσα ακούστηκαν ε, σήμερα για το θέμα της αφήνειας. Ίσως να επαναλάβω τα όσα είπε και η φίτριά μου πριν νωρίτερα, ότι δηλαδή ο κανονισμός βρίσκεται στην αρχή της διαδικασίας και υπάρχει ολόκληρο το κομμάτι της διαδικασίας και της εφαρμογής που επιτρέπει την εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τη, τα επίπεδα που θα συμφωνηθούν. Δεν θέλαμε εξ αρχής ε, στις Ρηξέλλες να ορίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και ίσως αν είναι καλό να θυμόμαστε ότι η, η, τα σώματα εφαρμογή, τα αρμόδια για την εφαρμογή θα είναι μαζί για να παρακολουθούν και να εξασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω και εγώ, όσο σαφέστερος είναι ένας κανονισμός, τόσο, όσο μ, σαφέστερα, σαφέστερη είναι οι ορισμοί, ε, τόσο λιγότερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στη φάση της αλληλοποίησης γιατί ακριβώς δεν, ε, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα της ερμηνείας. Να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε τι ήθελε να πει εδώ ο ποιητής νομοθέτης. Γι' αυτό και νομίζω ότι ε, κατά την νομοθετική διαδικασία για μας πρέπει να είναι πάντοτε ύψιστο στόχος να μην δημιουργούνται ποτέ και πουθενά παρεξηγήσεις. Χέλγα, ναι, συμφωνώ απόλυτα Υπάρχουν και κάποια προγράμματα όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή. Χρειάζονται ερμηνεία διάφορε διατάξει ή e-commerce για παράδειγμα. Εντάξει, δεν θέλω να ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα και να αρχίσουμε να το συζητάμε, αλλά το αναφέρω απλά για να δείξω ότι όταν υπάρχουν ασάφειε δημιουργούνται πολιτικά προβλήματα που κάποιοι μπορεί ενδεχομένω ορισμένε φορέ και να τα εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό και λέμε ότι όσο σαφέστεροι είναι ορισμοί τόσο καλύτερα και αυτό που είπε και η Σίλβια. Δεν θέλω να τα, να τα εντάξω όλα αυτά στην έκθεσή μου, τα έχετε όλα γράπτος. Η συνεργασία με τις οργανώσεις των νέων είναι ύψης της σημασίας και αυτό είναι το πνεύμα της έκθεσης μου γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί εμπειρογνώμονες και από αυτούς πρέπει να, αυτούς πρέπει να αφουγκραστούμε ε, και νομίζω ότι αυτοί είναι η βασική μας εταίροι, πλέον πολύτιμοι εταίροι μας, διότι γνωρίζουν τη δουλειά από κάτω, από τα μέσα. Αυτοί είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις δραστηριότητες με τους νέους και μπορούν να μας δώσουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες. Συγγνώμη, σε, δεν σε είχα δει. Ναι, ναι, πολύ σύντομα. Το ανοίγμα το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είναι κανονισμός, έχω αμφιβολία για το κατά πόσο θα το αφισβητήσουμε ή θα το θέσουμε. Η συμπαγή σε πολιτικές και νομικές βάσεις είναι απαραίτητες, όπως και οι οικονομικές, γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια προσπάθεια και εμεί είμαστε βεβαίω ε, διαθέσιμοι ως Επιτροπή για να αποσαφηνίσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να βάλουμε τα σωστά θεμέλια. Ήδη το βασικό ερώτημα μέσα στο Εράσμος ή εκτός Εράσμος δεν είναι και μικρό πρόβλημα και σε νομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Και το λέω βέβαια με πνεύμα συνεργασία αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι παρέμειναν ως το τέλος της συνεδρίασης εδώ στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ συνολικά για την εξαιρετική συνεδρίαση που είχαμε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου από τις 9 έως τις 12.30. Εώ τότε βεβαίω, θα έχουμε διάφορε ευκαιρίε να τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.